προσχώρησε στην ομάδα των φιλελευθέρων. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 4 κατέθεσε μια αιτιολογημένη γνώμη η οποία εάν ε, δεν ε, φέρουν αντίρρηση κάποιες ομάδες ή τουλάχιστον 40 συνάδελφοι τότε θα ε, προσθεθεί και αυτή στα πρακτικά της συνεδρίασης. Περνάμε κατόπιν συναρπαστικές ανακοινώσεις του Προέδρου. Σύμφωνα με το άρθρο 87α παράγραφος 6, ο Πρόεδρος της Διάσκεψης των Προέδρων Επιτροπών μου είπε πως δεν υπάρχει καμία αντίρρηση έναντι δύο συστάσεων